Äh, Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση που είχαμε αφήσει στη μέση το πρωί. Έχουμε ένα σημαντικό σημείο στην ημερήσια διάταξη. Είναι η παρουσίαση του προγράμματος εργασίας 2013 ε, του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Να καλωσορίσω και πάλι τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου, τον Βίτο Καλντέιρα, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας για το 2013 του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, κύριε Καλδέιρα, η ε, Επιτροπή Ελέγχου του Προπληκισμού είναι η δική σας επιτροπή, είναι η επιτροπή με την οποία συνεργάζεστε πολύ στενά. Βέβαια και οι υπόλοιπε επιτροπέ ε, ασχολούνται με τα αποτελέσματα των εκθέσεών σας. Ε, Βεβαίω ε, αυτό δεν είναι ένα καθήκον που αναλαμβάνουν μόνο οι ελεγκτές ας πούμε του προπολογισμού. Βεβαίω όλοι όσοι ασχολούνται με τα θέματα δαπανών μιλούν για χρηστή διαχείριση. Τη Δευτέρα είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον ε, Φανρομπαϊ, για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, αρκετά αντικρουόμενε απόψεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και πρέπει να, αυτό το πρόβλημα πρέπει να διευθετηθεί, πρέπει να λυθεί. Για τις υποχρεώσεις και για τις πληρωμές υπάρχει ένα κενό 50 δισεκατομμυρίων. Πρέπει να μιλήσουμε για καλύτερη δαπάνη, καλύτερη χρήση των κονδυλίων. Και αυτό βεβαίως είναι ίσως το βασικό καθήκον του ελεκτικού συνεδρίου. Να δει δηλαδή, να βρει πού υπάρχουν αδυναμίες, πού υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης και είμαστε βεβαίως εγγνώμονες στο ελεκτικό συνεδρίο για τη δουλειά που κάνει, αλλά και με ανυπομονησία περιμένουμε να μας πείτε τι έχετε ε, κάνει και τι προβλέπετε στο πρόγραμμα εργασίας σας για το 2013. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε και σας δίνω αμέσως το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα ευγενικά σας λόγια, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Κύριε τόρερ, θέλω να σας ευχαριστήσω, θέλω να ευχαριστήσω και την Επιτροπή σας που μου ξαναδίνετε τη δυνατότητα να σας μιλήσω σήμερα. Σήμερα με μεγάλη χαρά θα σας παρουσιάσω το τίσιο πρόγραμμα εργασίας ε, του συνεδρίου για το 2013 αλλά και τη στρατηγική μας μέχρι το 2017. Κατά την κατάρτιση της στρατηγικής και του προγράμματος εργασίας, ε, τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφελήθηκαν τα μάλα από τον επικοδομητικό διάλογο με τα μέλη της Επιτροπής σας, διότι είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε και διμερώς, αλλά και σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις και πραγματικά σας είμαι ευγνώμων ε, για γιατί μας δώσατε πολύτιμη συμβολή. Σήμερα τα θεσμικά όργανα που αντιπροσωπεύουμε παίζουν σημαντικούς και συμπληρωματικούς ρόλους για την εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής δημοκρατικής ευθύνης και λογοδοσίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο στόχος μας είναι τα δημόσια κονδύλια τα οποία διαθέτουμε να εκπληρώνουν τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης για να το πω απλά, στόχος ε, του συνεδρίου για τα επόμενα πέντε χρόνια είναι να συνεργαστεί στενά με το κοινοβούλιο, αυτό το κοινοβούλιο και το ε, τονίζω αυτό γιατί είναι φυσικό ότι δίνουμε προτεραιότητα στην δική σας επιτροπή. Το είπατε και εσείς κύριε ε, Πρόεδρε, γιατί είστε ο προνομιακός μας εταίρος εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά θα συνεργαστούμε και με οποιαδήποτε άλλη επιτροπή θελήσει να συζητήσει και να συνεργαστεί μαζί μας για τα πορίσματα των ελέγχων μας και των λογιστικών ασκήσεων. Αλλά βέβαια και με τους άλλους εταίρους θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε τη λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι είναι ε, στο επίκεντρο και της αποστολής μας. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι και ο καλύτερος δυνατός ε, τρόπος ε, να δώσουμε προστιθέμενη αξία για τους πολίτες μας στους καιρούς που ζούμε σήμερα, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας λογοδοσίας και των λογιστικών ελέγχων και γι' αυτό ε, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι συνεισφέρουν. Θα αναφέρω τρεις από αυτούς. Πρώτον, ότι ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καλούνται να στηρίξουν συντονισμένη δράση ε, των κρατών μελών εκτός του πλαισίου της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν παράλληλες δομές λογοδοσίας με πολύπλοκες διασυνδέσεις μεταξύ τους. Ένα παράδειγμα είναι για του λόγου του αληθές ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Δεύτερον, βλέπουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αναλαμβάνουν νέα καθήκοντα στο πλαίσιο τη νέα συνθήκη. Και αυτό έχει σημαντικέ επιπτώσει. Για παράδειγμα, ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του ενιαίου οπτικού μηχανισμού έθεσε για μια ακόμη φορά το ζήτημα της λογοδοσίας, της ευθύνης των κεντρικών τραπεζών αλλά και των χρηματοοικονομικών εποπτικών αρχών απέναντι στα κοινοβούλια και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Και τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερο χρησιμοποιεί μέσα πολιτικής, εργαλεία πολιτικής ε, που έχουν ως στόχο την προώθηση βιώσιμων δημοσίων οικονομικών, ανάπτυξης, θέσεων εργασίας, αλλά τα οποία δεν είναι εύκολο να ε, ελεγχθούν ε, δημόσια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα ρυθμιστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνήθως ε, δημιουργούν ε, κόστος εφαρμογής, το οποίο βαρύνει στις εθνικές αρχές ή τις επιχειρήσεις και απαιτείται και η κατάλληλη ρύθμιση για να μπορεί να αξιολογηθεί και ο αντίκτυπος αυτής εξ αρχής. Το ίδιο έχουμε κάποια δημοσιονομικά εργαλεία που χρησιμοποιούν δημόσια κονδύλια για τη μόχλευση των δημόσιων οικονομικών και τα οποία βγάζουν από τον ισολογισμό σημαντικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού και φυσικά πρέπει να υπάρχουν ειδικέ ρυθμίσεις ε, λογοδοσίας. Τέλο, έχουμε το πακέτο των προτάσεων που αφορούν το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτέ οι προτάσει θα επηρεάσουν σε πολλού τομεί πολιτική τη δημοσιονομική διαχείριση και κάποιες από αυτές τις αλλαγές θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά και την προσέγγιση του ελεκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά του συλλογιστικού ελέγχου. Με βάση όλα αυτά, λοιπόν, βασική προτεραιότητα του ελεκτικού συνεδρίου για την επόμενη πενταετία θα είναι να παράγουμε και να σα παράσχω προϊόντα τα οποία θα βελτιώσουν τη λογοδοσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δημόσια κονδύλια που θα πρέπει να διατεθούν για την επίτευξη των στόχων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει ω πρώτο βήμα να δούμε πού ε, κινδυνεύει περισσότερη λογοδοσία και χρηματοοικονομική διαχείριση. Και για αυτό το λόγο το 2013 το συνέδριο θα ετοιμάσει δύο αναθεωρήσεις, τοπίου όπως τις λέμε. Η μία θα αφορά τα ελλείμματα στον τομέα του λογιστικού ελέγχου και της δημόσιας λογοδοσίας και η δεύτερη την κάλυψη των κινδύνων, ε, των ρίσκων ε, στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Αυτού του είδους οι αξιολογήσεις και οι αναθεωρήσεις πιστεύουμε ότι είναι μία γνωμοδότηση κατά κάποιο τρόπο του συνεδρίου που δίνει μία γενική επισκόπηση των ζητημάτων που σχετίζονται με τα δημόσια οικονομικά που πρέπει πιστεύω να λάβουν υπόψη του οι χαράκτε πολιτική για την ανάπτυξη των προτάσεων. Θα συνεχίσουμε όμω να γνωμοδοτούμε και για συγκεκριμένε νομοθετικέ προτάσει, αφού βέβαια αυτέ καταρτιστούν, είτε κατόπιν ετήματο άλλων θεσμικών οργάνων, είτε και ιδέα πρωτοβουλία εφόσον θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν σκόπιμο. Για παράδειγμα, θα δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή στι νέε νομοθετικέ προτάσει για τον κανονισμό πλαίσιο για του εκτελεστικού οργανισμού, δυνάμει του άρθρου 208 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού. Το 2012 το συνέδριο έδωσε γνωμοδοτήσεις για πολλές από τις προτάσεις του νομοθετικού πακέτου για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το 2013. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στις διάφορες φάσεις, στάδια και επίπεδα της νομοθετικής διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά τώρα την ετήσια έκθεση του συνεδρίου για την ε, εφαρμογή, για την υλοποίηση του προπολογισμού της Ένωσης, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές, τους στόχους, τους κανόνες και τα ελεκτικά συστήματα που βλέπουμε να χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς πολιτικής μετά το 2013. Για το ε, οικονομικό έτος 2012 ε, έχουμε διατηρήσει τη δομή και την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης και θέλουμε να υπάρχει συγκρισιμότητα με τα προηγούμενα έτη στο τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο. Από την αρχή όμως του νέου δημοσιονομικού πλαίσιο, της νέας περίοδου προγραμματισμού, η προσέγγιση του συνεδρίου σε ό,τι αφορά τους λογιστικούς ελέγχους θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, ώστε να λάβουμε υπόψη οποιαδήποτε νέα πληροφορία και ε, διαβεβαιώσεις μας παρέχεται η Κομισιόν Εθνικές Αρχές στο πλαίσιο του στερικού ελέγχου. Ήδη προετοιμαζόμαστε για πανενδεχόμενο. Και ίσως αυτό μας οδηγήσει στο να επαναξιολογήσουμε και τη δομή των ειδικών εκτιμήσεων που παρέχουμε. Η προσέγγιση του συνεδρίου στην ετήσια αναφορά της Κομισιόν σε ό,τι αφορά τι επιδόσεις είναι ένας άλλο τομέα όπου αναμένουμε εξελίξεις. Είχαμε σημειώσει το Δεκέμβριο 2012 απαντώντα στη δεύτερη έκθεση εξολόγησης τη Κομισιόν δυνάμει το άρθρο 318 της Συνθήκης ότι θα πρέπει να τεθούν κάποια βασική ακρογωνή λύθη για μια αξιόπιστη διαχείριση των επιδόσεων και αξιόπιστο σύστημα αναφοράς. Και φυσικά η Κομισιόν μπορεί να διαβουλευτεί με το συνέδριο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Και στη συνέχεια, αφού πλέον θα έχει πονηθεί έκθεση, θα θεωρήσουμε κατά πόσον θα μπορούσαμε και εμείς τις πληροφορίες αυτής της έκθεσης αξιολόγησης να συμπεριλάβουμε στη δική μας ε, ε, ετήσια εργασία στο πλαίσιο του λογιστικού ελέγχου. Έρχομαι στις ειδικέ εκθέσεις. Θα επικεντρωθούμε σε ζητήματα που φαίνεται να χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο κινδύνου, δημόσιο ενδιαφέροντο ε, και δυναμικού για παροχή προστέμενη αξία. Θα κεντρωθούμε κυρίω σε θέματα επιδόσεων, απόδοση, ιδίω για την ανάπτυξη και την απασχόληση, την προστέμενη αξία, τα δημόσια οικονομικά, το περιβάλλον και τη δράση για την καταπολέμηση αλλαγή του κλίματο. Αυτέ οι προτεραιότητε αντικατοπτρίζονται ήδη σε μεγάλο βαθμό και στο φετινό ε, πρόγραμμα εργασία. Πράγματι, το ίμιση των 20 ειδικών εκθέσεων που προτιθέμεθα να δημοσιεύσουμε εντός του 2013 θα αφορούν τη βιώσιμη αηφόρο ανάπτυξη. Για παράδειγμα, οι δύο εκθέσεις οι οποίες δημοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο καλύπτουν επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και στη διαχείριση των δημοτικών ε, αποβλήτων τα σχετικά σχέδια υποδομή δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τώρα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, σχεδιάζουμε να δημοσιεύσουμε μια έκθεση εντός 2013 για την προστιθέμενη αξία στα γεωργικά προϊόντα ή προϊόντα δασοκομεία και θέλουμε επίση να εγκρίνουμε μια έκθεση για το χρηματοοικονομικό μέσο για το περιβάλλον. Το 2013 θα καλύψουμε με ελέγχου και τι εξωτερικέ δράσει σχέση με την Αίγυπτο, την Παλαιστινιακή Αρχή, την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την παροχή βοήθεια στην Κεντρική Ασία. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, απάντηση, την ανταπόκρισή μας στην δημοσιονομική κρίση, επεξεργαζόμαστε λογιστικούς ελέγχους για την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος και για τη διαχείριση ε, της, ε, του σωσίου πληρωμών και τη σχετική βοήθεια. Οι ειδικέ εκθέσεις του συνεδρίου περιλαμβάνουν πολλές συστάσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την απόδοση. Έτσι έχουν σχεδιαστεί Πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι αποδεκτέ και εφαρμόζονται. Αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στην όλη διαδικασία τη λογοδοσία. Το 2013 το συνέδριο θα δημοσιεύσει τη δεύτερη ειδική έκθεση follow-up, έκθεση παρακολούθηση, για να εστιάσουμε περισσότερο στι δράσει αντιμετώπιση ε, των στάσεων προηγούμενων ειδικών εκθέσεων και θα μελετήσουμε τα επιτευθέντα αποτελέσματα. Αν θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τη συμβολή μα στη λογοδοσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. θα πρέπει ω ελεγκτικό συνέδριο και να είμαστε, αλλά και να φαίνεται ότι είμαστε ένα οργανισμό ε, με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και υψηλή απόδοση. Γιατί έτσι μόνο θα εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία μα. Για να πετύχουμε στο στόχο αυτό σε ένα εξελισσόμενο, σε ένα μεταλλασσόμενο περιβάλλον ενωσιακό, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε ε, το συνέδριο και πιο γρήγορα και ταχύτερα. Την επόμενη πενταετία λοιπόν θα δώσουμε προτεραιότητα στα εξή. Πρώτα απ' όλα να αναπτύξουμε περισσότερο τον ε, οργανισμό μας σε ένα επαγγελματικό ελεγκτικό οργανισμό, να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία μας και επίσης να δείξουμε την απόδοση και την ε, λογοδοσία τη δική μας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει κάποιες σχετικές δραστηριότητες, παραδείγματο χάρη μια αξιολόγηση από ομοτήμους ε, των πρακτικών μας ε, στον τομέα του λογιστικού ελέγχου και θα ε, βασιστούμε και στις συστάσεις ε, της προηγούμενης τέτοιας αναφέρω ομοτίμου του 2008. Επίσης θέλουμε να εξορθολογήσουμε τις διεργασίες μας, τις διαδικασίες μας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των μετόχων μας και επίσης το, συγγνώμη, των ενδιαφερομένων μερών και βέβαια να μπορέσουμε να δώσουμε πιο ποιοτικές και έγκαιρες εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις. Με βοήθεια επίση εξωτερικού συμβούλου αναπτύσσουμε και την στρατηγική μα, τον των επικοινωνιών και των εξωτερικών σχέσεων και επικαιροποιούμε, ενημερώνουμε του βασικού δείκτε επιδόσεων που πρέπει να αναφέρονται στι ετήσιε εκθέσει δραστηριοτήτων μα για τα οικονομικά είτε από το 2013 και μετά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, τα επόμενα πέντε χρόνια το Ελεγκτικό Συνέδριο δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή σα, βέβαια, για να βελτιωθεί η λογοδοσία, η ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι πολίτε να είναι ήσυχοι ότι τα οικονομικά του συμφέροντα τη χάνουν προστασία και ότι τα χρήματά τους ε, αξιοποιούνται με σοφό τρόπο και σε συμμόρφωση με τους κανόνες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Äh, Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας σας. Έχουμε και τα έγγραφα βεβαίως που μας το παρουσιάζουν. Ευχαριστούμε που μας τα έχετε δώσει. Ευχαριστούμε και που μας το παρουσιάσατε. Το ελεγκτικό συνέδριο Νομίζω ότι έχει λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει ε, κατά καιρού στην ομάδα μας εδώ, στην ανταλλαγή ε, απόψεων που κάνουμε. Ε, νομίζω λοιπόν ότι είναι αρκετά επικοδομητική αυτή η συζήτηση και βεβαίως Χαίρομαι που ενδιαφέρεστε και εσείς για, την, ε, για τη δική μας την ε, δουλειά, για την... Ε, γιατί ούτως ή άλλως οι εκθέσεις σας πάντα δημιουργούν πολλά κίνητρα για συζήτηση. Και να πω επίσης ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον έγινε μια συζήτηση από μένα με τον αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Παγκόσμια Τράπεζα, είπε ότι στον λογιστικό έλεγχο ε, έχουν υπάρξει προβλήματα τυπικά για το ε, πώς προχώρησε το ελεκτικό συνέδριο με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θα είναι λοιπόν σημαντικό το θέμα αυτό γιατί ίσως ε, είμαστε ο δεύτερος ή ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος χρηματοδότησης παγκοσμίως. Και βεβαίως Πρέπει να δώσουμε λογαριασμό και στους ε, φορολογούμενους. Πρέπει να είμαστε διαφανείς. Αυτό είναι ένα σημείο που πραγματικά θα θέλαμε να το συζητήσουμε και εγώ ε, το σημείωσα πολύ θετικά ότι στο πρόγραμμα εργασίας σας, Πρόεδρε, Μιλήσατε για τις δαπάνες που εμπίπτουν στην αναπτυξιακή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν θέλω να προκαταλάβω τη συζήτηση. Έχω κι εγώ όμως να θέσω κάποια ερωτήματα, αλλά να δώσουμε και στα μέλη της Επιτροπής να πάρουν το λόγο. Πρώτος, ο κύριος Οντί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ονόματι της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα ήθελα να σας χαιρετήσω, κύριε Πρόεδρε Καλτέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη τη δουλειά που κάνετε επικεφαλής του σημαντικού αυτού θεσμού στον οποίο βασιζόμαστε. Και αν επιτρέπετε θα ήθελα να χαιρετήσω και την Λιάνα Ιβάνοβα που σας συνοδεύει ε, και που έμεινε για λίγο σε αυτό ε, το χώρο, ε, διορίστηκε την κυβέρνηση της και έχει την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου. Για το έγγραφο και για την παρουσίαση που κάνατε, για το έγγραφο θέλω να μιλήσω. Ο πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών που είναι δίπλα σας επέστησε την προσοχή σας στο ότι εμποδιζόμεθα λίγο εμείς οι βουλευτές από αυτό το θέμα που έθεσαν αρχικοί κρατών κυβερνήσεων να αφορά στους πληρωμών και πιστός υποχρεώσεων. Ο Επίτροπος μας είχε εξηγήσει ο Αρμόδιος ότι η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση θα είχε ένα έλλειμμα 9 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι Υπουργοί Οικονομικών, ανεξάρτητα από τη δυσκολία διαχείρισης των ε, δημοσιονομικών των κρατών, μας είπαν τα νέα δισεκατομμύρια δεν μπορούσαν να πληρωθούν. Είναι οφειλόμενοι οι λογαριασμοί. Πίσω από τα 9 δισεκατομμύρια υπάρχουν δικαιούχους. Και σε μια ήπειρο όπως η δική μας, να μην είμαστε ικανοί να τιμήσουμε τους λογαριασμούς, τα, ωφέλη ε, που αφορούσαν έργα ε, επιτόπου αφορούσαν το έρασμο στα ευρωπαϊκά ταμεία, ε, αφορά άτομα που υπέβαλαν ε, έργα και εγκρίθηκαν και δεν μπορεί να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να δώσουν τους πόρους. Σας το λέω αυτό διότι εμείς ανησυχούμε ως βουλευτές ε, και θα ήθελα να σας ρωτήσω μήπως θεωρείτε ότι το ελεκτικό συνέδριο θα μπορούσε να παίξει το ρόλο κάποιου φορέα που χτυπάει τον κόδον του κινδύνου. Αν η συνθήκη δεν γίνεται σεβαστή. Αν είναι, δεν είναι ισολογισμένοι οι προπολογισμοί μας, δεν μπορεί το ελεκτικό συνέδριο που παρακολουθεί να ειδοποιεί τους βουλευτές, τους υπουργούς και να λέει προσοχή θα σας λείψουν τελικά πριν το τέλος του χρόνου 10 δισεκατομμύρια πρέπει να βρείτε τους αναγκαίους πόρους αντί να γίνεται αυτό το θέαμα όπως έγινε πέρσι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου στο Όσλο είπε δεν υπογράφω όσο δεν έχω τη βεβαίωση ότι θα λάβω τα 9 δισεκατομμύρια και τελικά πήραμε τα 6 δισεκατομμύρια και 3 δισεκατομμύρια που τα παίρνουμε το 2013. Αυτό δεν προβάλλει μια καλή εικόνα. Νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο θα επιδεινωθεί διότι αρχή κρατών και κυβερνήσεων μας είπαν ότι θα υπάρξει διαφορά 50 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ ε, αναλήψη υποχρεώσεων και πληρωμών. Το ελεκτικό συνέδριο δεν μπορεί να είναι για μας μια, ένα είδος εξασφάλισης να παρακολουθεί τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενώσης καθημερινά και να παίζει το ρόλο αυτό κάποιου που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου υπάρχει το πρόβλημα. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μας πείτε για τις σχέσεις που έχετε με τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια και τους φορείς ελέγχου τους εθνικούς και καλές σχέσεις μπορείτε να δείτε ως τις περίπλοκες σχέσεις ε, με τα κράτη-μέλη και αν προχωρήσουμε προς ομοσπονδοποίηση θα έχουμε όχι πλέον διακυβερνητικές, θα έχουμε κοινοτικές σχέσεις, τόσο πάνω κάποιου του σχέσεις. Αυτή η συνεργασία ουσιαστικά πιστεύετε ότι θα κινηθεί ε, σε καλό επίπεδο πέρα από τη συνεργασία σε μεθοδικό επίπεδο. Το πρωί συζητήσαμε ε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είπαμε ότι χρειαζόμαστε ανεξάρτητο έλεγχο όσον αφορά τις οικονομίες που θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη-μέλη σε, σε διάφορα θέματα, σε διάφορους τομείς που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού, ε, χωρίς να, ε, να επηρεάζουμε την κυριαρχία. 27 ξεχωριστοί ε, στρατοί, εκατοντάδε ε, κτίρια σε όλο τον κόσμο που δεν μοιράζονται καν ένα φωτοτυπικό μηχάνημα. Όσον αφορά την πολιτική ανάπτυξη, σε Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη, έχουμε τα κράτη-μέλη, αυτά που κάνουν τα κράτη-μέλη, αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπω μπορεί να γίνει καλύτερο συντονισμό. Επιστημονική έρευνα, εντοπίσαμε 15-16 προγράμματα επί του δύο θέματος που χρηματοδοτούνται ασυντόνιστα. Θα δεχόσαστε το Ευρωπαϊκό Ελεκτή Συνέδριο μαζί με τους εθνικούς ελεγκτικούς φορείς να κάνουν ένα είδος ελέγχου όσον αφορά τις πιθανές εξοικονομήσεις. Να συντάσσετε έκθεση μεταφράσεως γλώσσας εργασίας να συζητείτε πολιτικά το θέμα στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δούμε τι οικονομίες θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Παίρνω και την ιδέα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας που ανήκει στην πολιτική μου οικογένεια που είπε εδώ και 15 μέρες οικονομίες ναι αλλά όχι εις βάρος ε, της οικονομίας. Μπορούμε να εξετάσουμε ό,τι οικονομία μπορούμε να καταφέρουμε να πετύχουμε θα μπορούσε να μας βοηθήσει να δώσει ένα χεράκι το ελεκτικό συνέδριο στον ρόλο που παίζει ή θα πρέπει να ζητήσει τη συνδρομή ενός εξωτερικού ελεκτικού φορέα. Θα ήταν κρίμα κάτι τέτοιο. Και κάτι άλλο, διότι μακρηγόρησε. Στην έκθεσή σας σελίδα 4 που αφορά το πρόγραμμα εργασιών αναφέρεστε εκτενώς τις αρμοδιότητες του ελεκτικού συνεδρίου, στις ε, γνώσεις θα ήθελα να αναφέρετε και ανεξαρτησία. Η λέξη ανεξαρτησία να αναφέρεται, διότι εμείς θέλουμε οι ελεγκτές να είναι ανεξάρτητοι και κάπου στη στρατηγική ή στο έγγραφο θα μπορούσατε να αναφέρετε αυτή την ανεξαρτησία. Και τελευταίο σημείο, μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερο όσον αφορά την αξιολόγηση από τους ομοτήμους. Ποιος δημιουργεί το σώμα που αξιολογεί το συνέδριο. Λίγα λόγια. Μπορείτε να μας πείτε εσείς που ελέγχετε, από ποιους ελέγχεστε. Ευχαριστώ. Άλλος. Κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Έχουμε λάβει αρκετές εκθέσεις σας αυτή τη χρονιά. Ας πούμε για τον σεισμό στην Άκουιλα. Ζητήσαμε να γίνουν οι λογιστικοί έλεγχοι στην Κομισιόν. Θέλαμε να μάθουμε την, ε, τις πληροφορίες από αυτό και πραγματικά περιμένουμε να μας υποβάλλετε τις σχετικές πληροφορίες. Θα ήθελα για την ειδική έκθεση για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων να κουβεντιάσουμε λίγο για το Foreign Policy Instrument γιατί μιλούμε για κονδύλια για την εξωτερική πολιτική και σημαντικό είναι στις δικές σας, ε, στο δικό σας σκεπτικό, ακριβώς για αυτά τα κονδύλια της ε, υπηρεσίας ε, εξωτερικών δράσεων να σας απασχολήσει το, το θέμα αυτό γιατί ούτως ή άλλως έχει πρόσβαση και η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων στα κονδύλια για την εξωτερική πολιτική. Άλλος κανείς? Όχι. Οπότε, Πρόεδρε, να κάνω εγώ δύο, να θέσω εγώ δύο ερωτήματα η Ίνγε έθεσε το θέμα της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων. Ένα θέμα που όταν συζητούσαμε με τον Επίτροπο Πίμπαλξ μας είχε απασχολήσει. Και μας απασχόλησε κυρίως το θέμα για τα κονδύλια για την αναπτυξιακή συνεργασία. Και στην ετήσια έκθεσή σας και εσείς λάβατε θέση από αυτού και νομίζω ότι και στο πρόγραμμα εργασίας 2013 αυτός ο τομέας θα παίξει σημαντικό ρόλο. Ένα ερώτημα που θέλω να κάνω είναι η αναφορά που γίνεται για το ότι κάποια κονδύλια σε, σε περιφέρειες που είναι σε κρίση δεν θα έπρεπε να αποδίδονται σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις που μπορεί να έχουν δεσμούς με τρομοκρατικές οργανώσεις. Ε, το παράδειγμα ήταν το Πακιστάν συγκεκριμένα, όπου σε κάποια ΜΜΕ έγινε, υπήρξαν και κάποιες κατηγορίες, κάποιες επικρίσεις, ότι αυτά τα κονδύλια μπορεί να χρησιμοποιηθούν με λάθος, τρόπο. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το άλλο ερώτημα που απασχόλησε την Επιτροπή μας είναι η στήριξη του πληθυσμού της Συρίας. Ένα μεγάλο ε, κομμάτι της, ε, των κονδυλίων πάνε στην Συριανή κυβέρνηση. Οι πολίτες όμως της Συρίας εποφελούνται από αυτά τα κονδύλια άνθρωποι που βρίσκονται τώρα σε μια εμπόλεμη κατάσταση και εσείς ως ελεκτικό συνέδριο θεωρείτε ότι υπάρχουν δυνατότητες για να παρέμβουμε σε αυτό κάπως. Μετά, παρουσίαση του Συμβουλίου. Στην ετήσια έκθεση μιλήσατε για το, κόστος, ε, για το διοικητικό κόστος ε, του Συμβουλίου και του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από κοινού. Εσείς ξέρετε ότι αποφασίζουμε για την, για την απαλλαγή του Συμβουλίου Υπάρχουν ε, κάποιε φωνέ που λένε ότι πρέπει να δούμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών ξεχωριστά. Οπότε ερώτημα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών στην ε, ε, έκθεσή σας γιατί είναι, θεωρούνται ένα όργανο ή έχουν μπει στο ίδιο κομμάτι, υπάρχει λόγος να γίνει ένας τέτοιος διαχωρισμός ή μήπω είναι αδύνατο να γίνει τέτοιος ε, διαχωρισμός. Ε, εντάξει, αν δεν μπορείτε να απαντήσετε μπορεί να είναι όντως αρκετά εξειδικευμένη ερώτηση, μπορείτε να μου απαντήσετε αργότερα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, ο κύριος Οντί θέλει να προσθέσει κάτι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διστάζω να ξαναπάρω το λόγο και μάλιστα μετά από εσά, αλλά θα ήθελα να πω ότι στη σελίδα 5 του εγγράφου για το πρόγραμμα εργασιών για το 2013 αναφέρεται ότι το ελεκτικό συνέδριο θα συντάξει δύο εκθέσει πανοραμικέ, σφαιρικέ όσον αφορά τον κίνδυνο για την οικονομική διαχείριση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και άλλη έκθεση όσον αφορά τις, τα ελλείμματα, τα ελεγκτικά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και τι υποχρεώσει να ληφθεί υπόψη. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η τίτλη που επελέγησαν για αυτές τις εκθέσεις. Δεν ξέρω αν ήταν χρήσιμο να πούμε ότι συντάσσουμε ε, ε, μια έκθεση για τις ελλείψεις του ελέγχου. Το να λέει ότι θα κάνει έλεγχο το, δικα... ελεκτικό συνέδριο, καλό. Αλλά να λέει ότι υπάρχουν ελλείψεις και προβλήματα, δεν είναι καλό. Θα γίνουν εκλογές του χρόνου ε, και όλοι οι αντιευρωπαϊστές θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα κένα. Εκ των προτέρων να λέτε ότι υπάρχουν ελλείψεις κλπ. Έτσι φιλικά θα να σας πω ότι ίσως δεν είναι σωστό να προδικάζετε το αποτέλεσμα, τα πορίσματα των εκθέσεων. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε. Είναι πολλά τα ερωτήματα και αρκετά διαφορετικά. Παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα όσο καλύτερα μπορώ. Βέβαια, για ορισμένα εξ αυτών φοβούμαι ότι δεν μπορώ να δώσω μια απλή ε, απάντηση, μια ευθεία απάντηση, αλλά με τα χαρά ε, είτε σε γραπτή μορφή, είτε κάποια, σε κάποια μεταγενέστερη ευκαιρία θα απαντήσω. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ντίκη για τα καλά του λόγια. Ξεκινώ με το πρώτο σημείο για την Παγκόσμια Τράπεζα. Θα ήθελα να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα στις 27 Φεβρουαρίου θα υποδεχθούμε μια αντιπροσωπεία από την Παγκοσμία Τράπεζα για να συζητήσουμε ακριβώς πόσο θα, πώς θα μπορέσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Είναι η Ένωση ο δεύτερος μεγαλύτερος ε, χορηγός, δωρητής προς την Παγκόσμια Τράπεζα και υπάρχει αυτή η ανάγκη να κάνουμε ε, ελέγχους λογιστικούς. Η Παγκόσμια Τράπεζα όμως έχει κάποιες πληροφορίες. Εμείς θα πρέπει να δούμε μαζί τους ε, πώς ρεαλιστικά μπορούμε να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Έχοντας δηλαδή γνώση όλων αυτών των πληροφοριών. Θα προσπαθήσουμε να εργαστούμε με διαφάνεια. Οι ελεγκτέ μας στον τομέα της βοήθειας για τις ανθρώπινες χώρες, για τους τομείς που χορηγείται βοήθεια, είναι τομείς που θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε με τον δέοντα τρόπο. Επίσης, είπατε κύριε Πρόεδρε, και η κυρία Γκρέσλε βέβαια, για την, ε, υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Από μια διαφορετική σκοπιά ο κύριος Οντί κάποια Θα ήθελα να τα συγκεράσω κάπως, αν μπορώ, να δώσω μια απάντηση συνολική. Εμείς με τα εθνικά ιδρύματα λογιστικού ελέγχου συνεργαζόμαστε ώστε να είμαστε σε θέση να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτό το οποίο ο κύριος Οντί θεωρεί παρά, παράξενο τίτλο για μια έκθεση το οποίο πανοραμική δεν μιλάμε όμως μόνο για τις μεθόδους. Θέλουμε να δούμε και σε ποιους τομείς θα μπορούσαμε να κάνουμε κοινή δουλειά. Και ένα από τα στοιχεία όπου εντοπίσαμε ότι υπάρχει ανάγκη οι φορείς ελέγχου να μιλήσουν ξεκάθαρα και να πούνε ότι υπάρχει θέμα λογοδοσίας και πρόβλημα, έλλειμμα, είναι η προληπτική εποπτεία. Είναι ε, κατά κάποιο τρόπο οι αρμοδιότητες οι οποίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά μετά πλέον εχωρούνται στο εθνικό επίπεδο. Αν δείτε τον κύκλο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, το six-pack, το two-pack, όλες αυτές οι προτάσεις ένα συμπεφωνημένο ήδη πλαίσιο, θα καταλάβετε ότι πρέπει, υπάρχει ανάγκη να δούμε ποιος είναι υπεύθυνο και υπόλογο γιατί και σε ποιο επίπεδο. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους ελεγκτέ, αλλά και το Εθνικά Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους εθνικούς Ελεγκτέ, το ε, ελεγκτικό συνέδριο, το ευρωπαϊκό κτλ. Για να απαντήσω λοιπόν στο ερώτημά σα. είμαστε διατεθειμένοι να εργαστούμε και ακόμη και πιο πέρα από αυτό το πλαίσιο και με του ομολόγου μου, προέδρου ε, των Εθνικών Αλληλεκτικών Συνεδρίων, έχω θέσει το θέμα αυτό για να δούμε αν υπάρχει ε, περιθώριο, γιατί δεν έχουμε και πολλού πόρου στη διάθεσή μα. και πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη μα και τι προτεραιότητε ε, των Εθνικών Αλληλεκτικών Συνεδρίων που μπορεί να μην συμφωνούν απόλυτα πάντοτε με τι δικέ μα προτεραιότητες. πώ μπορούμε όλα αυτά να τα συγκεράσουμε για να έχουμε μια κοινή διάσταση και να δούμε πού μπορούμε να εντοπίσουμε το που θα μπορούσαμε να έχουμε οικονομίες. Να εργαστούμε δηλαδή εκεί που πολλές φορές συμπίπτει το έργο μας στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, is... Θα ξεκινήσει ένας έλεγχος για το όργανο το οποίο είπατε που δεν είναι ακριβώς όργανο, τέλο πάντων, αλλά ε, έχουν ε, έχουμε οργανώσει αυτόν τον άλλο το είπε, αναφέρθηκε σε αυτό και η κυρία ο κύριος Στόιρ και ο κύριος Όντι. Δεν ξέρω αν θα δημοσιεύσουμε το 2013, αλλά ίσως στις αρχές του 2014 θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μια συνολική εικόνα της υπηρεσίας αυτής, της ΕΙΕΔ, που είναι ένα ιονή όργανο της Ένωσης. Και όλα αυτά βέβαια θα τα συσχετίσουμε και με το στοιχείο των ε, κτίριων και την πολιτική των κτίριων. Τώρα, οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί σε σχέση με τη βοήθεια, την ενίσχυση που παρέχει η Ένωση μέσω φορέων όπως ΜΚΟ και άλλοι. Βοήθεια λοιπόν που διεχτεύεται στι τρίτε χώρε ε, να εξασφαλίσουμε να μην φτάνει στα λάθο χέρια, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που ακούστηκε εδώ. Σύντομα θα έχουμε μια ε, έκθεση που θα δημοσιεύσουμε για έναν έλεγχο στην Αιγυπτό και για την Παλαιστινική Αρχή, επίκειτη δημοσίευση. Σημειώνω τι ανησυχίε σα για τη Συρία. 2013 και για την Κεντρική Ασία ε, σκοπεύουμε να δημοσιεύσουμε μία έκθεση σε σχέση με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ανησυχίες. Αυτά σε ό,τι αφορά την κάλυψη του πολύ σημαντικού αυτού τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της αναπτυξιακής βοήθειας και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στο πέσο των νέων της αρμοδιοτήτων. Όλα αυτά είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας και νομίζω ότι ανταποκρινόμαστε στις ανησυχίες σας. σημείωσα όσα είπατε και θα προσπαθήσω να τα συμπεριλάβω βέβαια στο μελλοντικό μας έργο χωρίς να σας υπόσχομαι ότι το 2013 θα έχουμε έκθεση για όλα αυτά τα θέματα. Θέλω να είμαι ειλικρινής, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα φροντίσουμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα και να διασκεδάσουμε τις ανησυχίες σας στους τομείς αυτούς. Ένα άλλο ερώτημα Είχε να κάνει με το Συμβούλιο. Γιατί δεν διακρίνω μεταξύ Συμβουλίου αφενός και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αφετέρου. Εμείς ελέγχουμε τον προπολογισμό. Πρώτα πρέπει να δούμε πώς στον προπολογισμό θα ορίζεται ξεκάθαρα τι πηγαίνει στο κάθε ένα από τα δύο όργανα. Θα το επεξεργαστούμε και ίσω και διμερώς θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τις δικέ σα ανησυχίε για να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να ανταποκριθούμε. Πάντως πρέπει να σας πω ότι κάθε χρόνο στου ετήσιους μας ελέγχου εξετάζουμε αυτό το όργανο και αν υπάρχουν διαφορές σε οριζόντια θέματα, εκεί κάνουμε το διαχωρισμό μεταξύ των δύο. σε ό,τι αφορά τα προβλήματα τα οικονομικά και για το νομισματικό πλαίσιο αλλά και για το τρέχον πλαίσιο και αν μπορεί το συνέδριο να δραματίσει ένα διαφορετικό ρόλο να προειδοποιεί, να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, θέλετε. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το κάνει ήδη το Ελληνικό Συνέδριο εδώ και κάποια χρόνια και αρκεί να διαβάσετε την ετήσια έκδοση του 2011 τη συζητήσατε χθε νομίζω. Ήδη εκεί λέμε το 2011 το ίδιο πρόβλημα ανέκυψε και θα μπορούσαμε να είχαμε 5 δις εάν πιστώσεις πληρωμών είχαν καλυφθεί με τα βάρυτα κονδύλια. Δύο προβλήματα έχουμε. Το πρώτο είναι ότι έχουμε μια ατυπική περίοδο υπό την έννοια ότι πλήττονται από την κρίση. Τα κρατημελιάρια εθνική χρηματοδότηση παρουσιάζει καθυστέρηση, πλησιάζουν στο τέλος περίοδου και υπάρχουν μεγάλες πιέσεις να εκταμιευθούν τα χρήματα, να γίνουν οι πληρωμές. Και εκεί έχουμε το θέμα με τις αναλήψεις υποχρεώσεων, τα commitments. Όταν τα κράτη-μέλη λοιπόν κάνουν τον προγραμματισμό τους, τον προγραμματισμό τους για τι πληρωμέ. φτάνουν στο τέλος του έτους, αλλά δεν έχει γίνει μια σαφής πρόβλεψη για όλο το χρόνο, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει καθαρά πρόβλημα με τον προγραμματισμό και με την ε, διάθεση και πρόβλεψη των πόρων. Οι χώρες που έχουν ανάγκη λοιπόν από πιστός πληρωμών θα πρέπει να επεξεργαστούν ε, πολύ πιο καλά τα στοιχεία για να μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα ταμιακά διαθέσιμα. Διότι ένα μέρος των πιστώσεων πληρωμών φτάνει στο, τρίτο, στο τέταρτο συγγνώμη, τρίμηνο του έτους και ακόμη κι αν εμείς καθημερινά από πλευρά ελεκτρικού συνεδρίου παρακολουθούμε και επιβλέπουμε τα πράγματα, ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επομένως, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εδώ και χρόνια είναι να κρούμε το, να με το συναγερμό αν θέλετε. Αλλά υπάρχει ζήτημα προγραμματισμού και πρόβλεψης. Πρέπει να είναι πιο καλή η πρόβλεψη, η πρόγνωση από πλευράς κρατών μελών. Και οι πληρωμές θα πρέπει κάπως να εξαπλώνονται χρονικά, να μην φτάνουν όλες τον ίδιο μήνα, ώστε τα κράτη-μέλη που υπόκεινται σε σημαντικές ε, δημοσιονομικές και αταμικές πιέσεις να μπορούν να αποκριθούν στα αιτήματα ε, πληρωμών. Αν προβλέψουμε ήδη τώρα ένα γενικό δημοσιονομικό πλαίσιο που παρουσιάζει μεγάλη διαφορά μεταξύ των ε, πληρωμών και των ανλήψεων υποχρεώσεων, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όταν θα κάνουμε τις προβλέψεις για τις πιστώσεις πληρωμών για όλο το έτος. Και θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 ξεκίνησε με καθυστέρηση. Για δύο χρόνια δεν έγιναν σχεδόν καθόλου πληρωμές. Ξεπιστοποίηση των εθνικών συστημάτων, των αρμόδιων εθνικών αρχών. Έπειτα μας χτύπησε η κρίση και καθυστερήσαμε με την έναρξη των προγραμμάτων. Τώρα λοιπόν πλησιάζει το τέλος αυτής της περίοδου προγραμματισμού και είναι η ώρα να γίνουν οι πληρωμές. Και ο πιο σημαντικό συναγερμό, αν θέλετε, που μπορούμε να σημάνουμε ω ελεκτικό συνέδριο είναι να υπενθυμίζουμε κάθε στιγμή, κάθε χρονιά, τις λεγόμενες ε, υπνότουσες ε, αναλήψεις υποχρεώσεων, δηλαδή το υπόλοιπο προσεκαθάριση. Εκεί βλέπετε τη διάσταση αυτή η οποία χτυπά την πόρτα θέλετε, για, το, για την περίοδο 2007-2013. Δηλαδή, κονδύλια που έχουν δεσμευθεί υπάρχει νομική δέσμευση και δεν έχουν εκταμιευθεί ακόμη. Για το 2011 περιμένουμε να έχουμε κάποιες, ε, κάποια νούμερα για να έχουμε τον ετσιού προπλησμό της Ένωσης. Μιλάμε για τρία χρόνια πληρωμών αν ε, παραμείνει ο ρυθμός ο σημερινός. Και έτσι θα έχουμε προβλήματα. Το βλέπουμε από τώρα ε, με τα ταμιακά διαθέσιμα. Άρα έχουμε αυτά τα προβλήματα και με το υπόλοιπο που σε καθάρισε, επαναλαμβάνω. Θα μπορούσε, επομένως, ε, το ελεκτικό συνεδρίο να σημαίνει συναγερμό και το κάνει ήδη, θα μπορούσαμε ίσως να επιμείνουμε ακόμη περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει και αυτή να αναλάβει τις ευθύνες της θα πρέπει να φροντίσει όλες τις δημοσιονομικές προβλέψεις, οι ανάγκες ε, για πιστώσεις ε, στη διάρκεια του έτους, αλλά και στο τέλος του έτους να είναι ρεαλιστικές. Τώρα, η ανεξαρτησία του ελληνικού συνεδρίου. Μπορεί να μην το αναφέρουμε ρητά στο πρόγραμμα εργασίας, το αναφέρουμε όμως ε, στο έγγραφο στρατηγικής. λέμε ότι είναι στο DNA μας, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Δεν αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά ε, το ελεγκτικό συνέδριο, παρά ως έναν ανεξάρτητο οργανισμό και φορέα. Αυτό το επιβάλλει και η συνθήκη και το δείχνει και η καθημερινή πρακτική, πιστεύω. Και θα είμαι πάντοτε ε, ένας από τους περασπιστές της ανεξαρτησίας αυτής. Σας ευχαριστώ πάντως που το αναφέρετε και σίγουρα θα λάβουμε τα σχολεία σας υπόψη. Τώρα, πού βρισκόμαστε στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης από Νοτίμου. στο peer review, έχει ξεκινήσει. Έχουμε μια ομάδα την οποία αποτελούν ε, ομότιμοι από το Γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι ο Γενικός Ελεγκτής ε, της ε, Σουηδίας και εκπροσωπείται και το Γερμανικό Ελεγκτικό Συνέδριο, ας πούμε ο Γενικός Προϊστάμενος, οι οποίοι εδώ και κάποιους μήνες, από τον Νοέμβρη συγκεκριμένα, μελετούν όλους τους απαραίτητους φακέλους και περιμένουμε να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους εντός του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Άρα, φέτος θα δημοσιευτεί η τελική έκθεση και βέβαια θα σας ενημερώσουμε σε αυτό το χρόνο για τα αποτελέσματα αυτής της αξιόλογης από ομοτήμους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που οι τρεις αυτοί τόσο σημαντικοί φορείς με τόσο μεγάλο κύρος δέχτηκαν να κάνουν την αναθεώρηση από ομοτήμους. Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολευτήκαμε να βρούμε ομοτήμους, γιατί είναι πολύ του σειρμού από τη μια πλευρά. Υπάρχουν πολλά αιτήματα, αλλά γίνεται δωρεάν από την άλλη πλευρά. Πληρώνουμε δηλαδή έξοδα μετακίνηση. Θα έχετε δει ίσω στον προπολογισμό μας ότι έχουμε μια κατηγορία που προβλέπει την ε, επιστροφή εξόδων μετακίνηση, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι ιδίες δαπάνες αυτών των φορέων που δέχονται να κάνουν την αξιολόγηση από ομοτήμους και χαιρόμαστε πάρα πολύ που προσφέρθηκαν οι τρεις αυτοί φορείς για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ε, τώρα, επειδή με ρωτήσατε γιατί διαλέξαμε αυτό τον ε, τίτλο, Public Deficits or Audit Deficits, αυτό το, το τίτλο που μιλάει για ελλείμματα ή ελλείψεις στον τομέα της λογοδοσίας και των οριστικών ελέγχων. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό το ελληνικτικό συνέδριο να μπορεί να κάνει μία ως το δυνατόν πιο διεξοδική δουλειά. Να μελετά όλες τις εξελίξεις και να βλέπει ακριβώς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αν όλα τα νέα εργαλεία και μέσα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Προληπτική εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. μέτρα για απόδοση λογαριασμών και λογιστικό έλεγχο όλων αυτών των λεγόμενων trust funds και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών. Μετά την έκδοση του Μεσαίου οργανισμού είχαμε κάποιες εξελίξεις ε, και έχουμε αναφέρει και κάποιες ε, ανησυχίες μας. Έχουμε εκφράσει απόψεις μας για τις προτάσεις αυτές. Και βέβαια θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει μια χαρτογράφηση όλων αυτών εμείς θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε αυτή τη γενική χαρτογράφηση, έναν άτλαντα ε, με όλες αυτές τις εξελίξεις για να δούμε ε, και επίσης να δούμε πού εντοπίζουμε εμείς πρόβλημα. Θα το επισημαίνουμε. Το είπαμε πολλές φορές και στην Επιτροπή σας και το έχετε πει και εσείς ότι το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό κάποιες φορές παραγωνίστηκε Και μα λένε κάποια εθνικά κοινοβούλια ότι δεν έχουμε κάτι εθνική κυριαρχία να εγκρίνουμε τον εθνικό μα προπολογισμό γιατί την δημοσιονομική πολιτική των κρατών μελών την ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι λίγο υπερβολικό μεν, αλλά δείχνει δε την ανησυχία που υπάρχει σε ό,τι αφορά την απόδοση λογαριασμών. Αν υπάρχει δηλαδή δημόσιος έλεγχος και αν μπορεί και αν έχει κάποιο ρόλο ο ελεγκτής εδώ για να διευκολύνει τα πράγματα. Έχετε λοιπόν ε, ζητήσει πολλές φορές να κάνουμε κάποιες εργασίες. Ορίστε εδώ ε, λέω ότι υπάρχουν κάποια ελλείμματα, υπάρχουν ελλείψεις. για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα. Γιατί να μην γίνει ένα έλεγχο εκεί, ποιο ελέγχει. Ποιος ελέγχει επίσης αυτό το μέσο την διευκόλυνση για τις εγγύσεις και τα δάνεια που έχει εσωματωθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Σίγουρα είναι σαφές ότι υπάρχει ε, έλλειμμα ε, δημόσιο ελέγχου. Γι' αυτό λοιπόν επιλέξαμε αυτό το τίτλο και ελπίζουμε με κάθε ταπεινότητα μέσα στο 2013 να μπορέσουμε να προβούμε στη χαρτογράφηση ε, ώστε να το πιο ξεκάθαρη χαρτογράφηση, όλα αυτά τα στοιχεία ακριβώς για να μπορούν οι νομοθέτες να στοχεύσουν καλύτερα τις διάφορες πτυχές ε, και να βρουν ικανοποιητικέ λύσεις. Και επιπλέον στο Σύνταγμα τη της Ευρωπαϊκής Ενώσης κάνουμε μια εξέλιξη εκτός συνθήκων. Έχουμε εξέλιξη εκτός συνθήκων. Έχουμε διάφορα μέσα, χρηματοπιστωτικό και άλλα, που δεν εμπνέονται από τη συνθήκη και το ελεγκτικό συνέδριο, το ευρωπαϊκό, είναι ένα θεσμικό όργανο που βασίζεται επί των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ούτως ώστε να εντοπίσουμε ακριβώς την προσέγγιση που χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι κάλυψα και το ερώτημα της κυρίας Γκρέσλε που αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, σε έναν έλεγχο που έχει ήδη δρομολογηθεί, θα το καλύψουμε αυτό και ελπίζω ότι η έκθεση για την Άκουιλα και το Αμπρούτσο ε, είναι κάτι που θα δημοσιευτεί αυτή την εβδομάδα. Εξάλλου, ένας, από ένα συνάδελφο πρώην μέλος της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Yeah, εγώ ευχαριστώ. Λεπτομερέστατες οι απαντήσεις σας στα ερωτήματα που σας έθεσαν. Ο κύριος Οντί θέλει πάλι το λόγο. Παρακαλώ. Όσον αφορά αυτή την πρόταση για το συναγερμό, είδα την παράγραφο, ξέρετε, την έκθεση του 2011 που έπρεπε να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο μήνα Οκτώβριο έτους 2012 και συζητήσαμε με πολιτικό στο θέμα το Φεβρουάριο του 2003, εγώ θέλω να μειωθούν όλες αυτές οι, προ... οι χρονικές προδιαγραφές. Εγώ ήθελα να επαγρυπνείτε διαρκώς αυτό, σε αυτό αναφερόμενο, αλλά σωστά το λέτε, αναφέρετε εδώ. Ευχαριστώ. Φτάσαμε στο τέλος του καταλόγου των ομιλητών. Οπότε το μόνο που μου απομένει, κύριε Πρόεδρε, είναι να σας ευχαριστήσω. Πάντα χαιρόμαστε όταν τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου είναι διατεθειμένα να μας απαντήσουν στις ερωτήσεις μας. Ε, ε, ούτως ή άλλως ε, και η εκθέση σας είναι βάση για, τις δικές μας, για τη δική μας εργασία. Ούτως ή άλλως ε, ε, αυτές είναι, ε, ένα από, είναι, αυτό είναι ένα από τα λίγα όργανα που έχει το Κοινοβούλιο ώστε να μπορέσει να αξιολογήσει ότι όντως γίνεται χρηστή διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων. Ούτως ή άλλως λίγες ευκαιρίες έχουμε να παρέμβουμε και να παρακολουθήσουμε τα οικονομικές δραστηριότητες. πάντα λαμβάνουμε ε, επιστολές, email, ε, μας έρχονται και μας μιλούν στους, ε, στις διάφορες εκδηλώσεις για το τι γίνεται με τα δημόσια οικονομικά. Πάντα υπάρχει φόβος από τους φορολογούμενους για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, τι γίνεται με τον προϋπολογισμό. Γι' αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να δώσουμε και θεσμικές εγγυήσεις και να εξασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια χρησιμοποιούνται με τον καταλληλότερο δυνατό τρόπο. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη δουλειά που έχετε να κάνετε στο έτος αυτό που τρέχει. Σίγουρα και τα κρατη αλλά και η Κομισιόν θα, με τη δική σας τη βοήθεια θα φροντίσουν ώστε να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια σωστά. Βεβαίως υπάρχει στενή συνεργασία και το είπατε και εσείς με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Και επίσης ε, ε, χαίρομαι που είπατε ότι θα, θα ε, επικεντρωθείτε κυρίως στους ελέγχους για τις επιδόσεις. Αυτό είναι όντως πολύ καλό. Και βέβαια τίθεται και το ερώτημα σε σχέση με το ευρωπαϊκό εξάμεινο για τον, για τον έλεγχο το δημοσιονομικό, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα εργαλεία που έχουμε, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι έχουμε κάνει αρκετά, μεγάλο, αρκετά μεγάλη απόσταση. Βεβαίως πάντα υπάρχει ανάγκη για να προχωρήσουμε περισσότερο. Και θα ήθελα να σας πω ότι ε, υπάρχει μια διακοινοβουλευτική διάσκεψη με τις επιτροπές που είναι υπεύθυνε για τον, κοινοβουλευτικό, ε, για τον ε, δημοσιονομικό έλεγχο από τα κράτη-μέλη. Και πραγματικά θα χαιρόμασταν πολύ αν και το ελεγκτικό συνέδριο μπορούσε να συμμετάσχει σε μια τέτοια συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας σας, εξ ονόματος όλης της Επιτροπής και βεβαίως ε, προσβλέπουμε στη μελλοντική συνεργασία μας. Συνάδελφοι, φτάσαμε στο τέλος της ημερήσιας διάταξης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στο διάφορα. Εγώ δεν έχω να θέσω κάτι. Οπότε να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ τη Γραμματεία. Ευχαριστώ το Ελεκτικό Συνέδριο. Ευχαριστώ το Ινκομισιόν, τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Ο Πρόεδρος ευχαριστεί και τους Δερμηνείς. Και εμείς τον ευχαριστούμε μπορούμε να κλείσουμε τη συνεδρίασή μας. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι 21 Φεβρουαρίου του τρέχοντος στις 9 το πρωί. Έτσι δεν είναι. 9 το πρωί. Θα τα πούμε την επόμενη φορά λοιπόν. Καλώς σας απόγευμα.